Συνάδελφοι, πέρασε η ώρα. Να ψηφίσουμε. Γιατί έχουμε και άλλα μολομέλειες, αντιπροσωπείες, ομάδες. Σημείο 1 της ημερησιάς μας, εγκρίνουμε την ημερήσια, δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις της Προέδρου, δεν έχω ανακοινώσεις. Σημείο 3. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αυτό 53. Ευαίσθητη νομοθεσία, πολλές συζητήσει. Είχαμε τον εισηγητή τον κύριο Βαρινέν ο οποίος νομίζω πρέπει να πάρει το λόγο παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, σύντομα επειδή έχουμε διάφορες συναντήσεις των σκιωδών. Ξέρετε, νομίζω όλοι σας τις θέσεις των διαφορών πολιτικών ομάδων. Να πω ότι γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, λυπάμαι που η Επιτροπή μας δεν μπορεί να λάβει μια ισχυρή θέση πολιτικής. Καταλαβαίνω ότι στην άφετη ενδεχομένω υπάρχουν αποκλήσει απόψεων κλπ. Αλλά η θα έπρεπε να σε θέση να έχει μια θέση ισχυρή όσον αφορά την πολιτική αυτή. Κάποιοι ίσως να νομίζετε ότι αν αποκλείσουμε το ECI τη χρηματοδότηση θα ήταν σημαντικό. Δεν θεωρώ όμως ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο να έχουμε αυτή την, ε, αυτό το capacity building τη σημασία που έχει η φύση του. Δηλαδή πώς γίνεται να έχουμε ανάπτυξη όταν οι κανόνες της πολιτικής ανάπτυξη δεν εφαρμόζονται από την αρχή και πώς θα μπορούσε η νομική βάση να επιτρέψει την ανάπτυξη αν οι ίδιοι οι κανόνες της ανάπτυξη δεν εφαρμόζονται. Αυτό για μένα είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Αν λοιπόν το αποτέλεσμα σημαίνει ότι αυτό το capability, αυτή η δυνατότητα δεν, δεν περιλαμβάνεται, τότε σημαίνει ότι για τις δικές μου τροπολογίες 1 και 4 θα πρέπει να τις καταψηφίσω στην τελική ψηφοφορία και θα πρέπει να αποσύρω το ίδιο μου το όνομα από αυτή την έκθεση. Αυτή είναι η δικιά μου τελική και ανυποχώρητη θέση. Αλλά ξέρω εκ των προτέρων ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γι' αυτό το λέω, και θα ήθελα να το πω αυτό ευθύ εξ αρχή, ξεκάθαρα. Ωραία, λέει πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Προτείνω να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα, γιατί είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι στην προηγούμενη ψηφοφορία. Κάνουμε μια δοκιμαστική πρώτα, έτσι, συνάδελφοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Μήπως κάποιος μπάσατε το κουμπί. Ψηφίσατε όλοι. Ναι, ιού. Ψηφίστε. Δοκιμάζουμε. Γιατί πριν είχαμε ένα πρόβλημα, ξαναλέω. Ναι, κάποιος μπορεί να ξέρει την κάρτα του μέσα στο μηχάνημα. Πέρας. Λειτουργεί. Τέλεια. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την κανονική ψηφοφορία τώρα. Και αρχίζουμε. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 43 και 44 μαζί. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 46. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Περάς. Εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ Οι 47 και 49 ήταν μαζί συγγνώμη λέει πρόεδρος συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αλλά οι σοσιαλιστέ να μου δείξουν πιο ξεκάθαρα την ψήφο, ε, γιατί δεν καταλάβουμε ακριβώ τι κάνουν. Συμβαστική δύο, λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. Ψηφίζετε όλοι, περάς, εγκρίνεται. Παρακαλώ, αναμάδα, δείξτε μας ξεκάθαρα τι ψηφίζετε. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά να σας βλέπουμε για να τελειώνουμε πιο γρήγορα. 51. Καταπίπτει και αυτή, οπότε πάμε στη συμβαστική 4. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. 53 ξαναλέει πρόεδρος, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 53. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Συμβαστική 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πάλι για τη συμβαστική 1. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολόγια 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 αποσύρθηκε. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενη πίπτη οπότε πάμε στην 56, λέει πρόεδρος. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το 57 άρχεται για το 57 ψήφισατε όλοι περάς εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ 64-65 μαζί διορθώνει τώρα πρόοδο υπέρ κατά αποχέ απορρίπτώνται. 66 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 71 71-72-73 μαζί. 71-72-73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 71-72 και 73. Νομίζω έχει περάσει, αλλά τέλο πάντων το ελέγξουμε. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται, ναι. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για την 75. Άρχεται η ψηφοφορία για την 75. Ψήφισατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές λέει πρόεδρος απορρίπτεται, απορρίπτεται, απορρίπτεται συγγνώμη λέει πρόεδρος να στους σοσιαλιστές 79 υπέρ κατά αποχές θα το κοιτάξουμε γιατί δεν είναι ξεκάθαρο λοιπόν Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι πέρας. Νομίζω εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. Τώρα αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δηλαδή εγκρίνεται διορθώνει η πρόεδρος. Ναι, ναι. Εγκρίνεται η συμβαστική 5, λάθος έκανα. Και περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 28. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 και 30 και 31 μαζί υπέρ κατά 29, 30 και 31, όλες μαζί αυτές. 25, because 5 was carried and those, those ones... Αφού εγκρίθηκε η συμβιβαστική 5, καλύπτονται ή καταπίπτουν. Και πάμε στην 28 τώρα. Την ψηφίσαμε. 29, 30, 31. Το καταλάβαμε. Ωραία. Προχωρούμε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 33 αρχίζει τώρα ηλεκτρονική επαλήθευση. Πήγα και τελειώνει. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ποια ήταν αυτή, οι δύο αλλά και κάποιες άλλες μαζί. Μάλιστα. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 41 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε σε αιτιολογικές αναφορές τώρα. Οι τροπολογίες 8, 9 και 7 μαζί. Όχι. Ο κύριος Κοράου. Πρόεδρε, ε, μια τεχνική διόρθωση προτείνω ε, στην 8, 9 και 7 νομίζω να πάνε σε τελογικές σκέψεις, recitals, όχι στις αναφορές στο citations, να πάει στα recitals. Γιατί αλλιώς θα υπήρχε τεχνικό, ε, βασικά νομικό πρόβλημα. Μάλιστα, αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ λέω και σκοράω. Πολύ ωραία, πάμε ψήφι υπέρ αυτών των τροπολογιών στα recitals. Υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Οπότε τώρα θα πάμε στην τροπολογία 10, ψήφι υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Η 11 κατά πίπτη και μπορούμε να ψηφίσουμε το σχέδιο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα ονομαστικά η ψηφοφορία. Vote Εγκρίθηκε 13 ψήφοι υπέρ 8 κατά και μία αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βάιρινεν. Φαντάζομαι τι θέλετε να πείτε. Ναι, κυρία Πρόεδρε, αποσύρω το όνομά μου από την παρούσα έκθεση. Να το αναλάβει κάποιο άλλο γιατί είναι ορφανή τώρα. Ψάχνουμε διαπραγματευτή. Μάλλον μου πέφτει με ένα κλήρο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό και θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ και τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε και τη γραμματεία. Πολύ ταχεία η διεκπαιρέωση